Στην έναρξη της προηγούμενης ε, συνόδου, η Επιτροπή Θεσμικών Υποθέσεων ε, πρότεινε μια ερμηνεία του παρατήματος 16 παραγράφου 1. Ε, εάν δεν υπάρχει κάποια αντίθεση σε αυτήν την ερμηνεία, βάσει του άρθρου 226 παραγράφου 3, δεν έχει λοιπόν ληφθεί καμία αντίθεση, επομένως θεωρείται ότι έχει εγκριθεί αυτή η ερμηνεία. Οι αρμόδιες επιτροπές έχουν διαβιβάσει δύο ορθωτικά σε τέσσερα κείμενα που ενεκρίθη το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βάσει του άρθρου 231 παράγραφος 4. Αυτά τα, αυτές οι, δια, διορθώσεις θα θεωρηθούν ότι έχουν εγκριθεί εάν σε, σε επόμενε 24 ώρες μια πολιτική ομάδα ή τουλάχιστον 40 βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν ζητήσουν να ψηφιστούν. Είναι διαθέσιμα και στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και θα αναφερθούν και στα πρακτικά της τρέχουσα συνεδρίασης. Την Τετάρτη, βάσει του άρθρου 78 του κανονισμού μαζί με τον πρόεδρο του Συμβουλίου ενεκρίθησαν 12 νομικές πράξεις της, της ε, κανονικής νομοθετικής διαδικασίας. Θα, δια, θα, θα δημοσιευτούν μαζί με τις, τα πρακτικά της σημερινής συνεδρίας αυτές οι 12 πράξεις. έχουμε λοιπόν στη σημερινή ημερήσια διάταξη βάσει του άρθρου 149 της ημερήσιας διάταξης ενέκριναν ε, οι πρόεδροι των πολιτικών ομάδων το σχέδιο οριστικής ε, ημέρησης διάταξης. Θέλετε